Κοινοβουλίου, τον κύριο Μάρτιν Σούλτς. Ο κύριος Σούλτς είναι γνωστός σε όλους μας για την σοβαρότητα, συνέπεια και επιμονή με την οποία υποστήριζε επί πολλά χρόνια τόσο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και ευρύτερα τις θέσεις του για μια Ευρώπη που πρέπει να κινείται σε προοδευτική κατεύθυνση και να ανταποκρίνεται στις ελπίδες των πολιτών της. Κύριε Πρόεδρε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, χαίρομαι που ανταποκριθήκατε αμέσως την πρόσκλησή μου να έρθετε στην Αθήνα και να απευθυνθείτε εδώ σε αυτό το χώρο στη Βουλή των Ελλήνων στους Έλληνες βουλευτές εδώ σε αυτόν τον τόπο που πριν από 2.500 χρόνια γέννησε τη δημοκρατία. Η επίσκεψή σας αυτή πραγματοποιείται σε μια περίοδο ιδιαίτερα κρίσιμη για την Ελλάδα, για την Ευρωζώνη αλλά και ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα, κύριε Πρόεδρε, καταβάλει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια να εξηγιάνει τα οικονομικά της και προωθεί πλήθος διαρθρωτικών αλλαγών. Η τεράστια αυτή προσπάθεια δεν είναι μόνο της κυβέρνησης, δεν είναι μόνο του Κοινοβουλίου, αλλά είναι κυρίως του ελληνικού λαού που υφίσταται μεγάλες και οδυνηρές θυσίες. Θα μου επιτρέψετε στο σημείο αυτό να θυμίσω ότι η Ελλάδα μέσα σε δύο χρόνια μείωσε το έλλειμμα του προϋπολογισμού κατά 6,5% το ακαθάριστο εγχώριο προϊόντος, κάνοντας τεράστιες προσπάθειες, τεράστιες περικοπές. Για να κάνω μια σύγκριση, όπως είπα και πρόσφατα στο Βερολίνο, όταν ενημέρωνα 100 βουλευτές του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος αλλά και του S5, για να κάνω μια σύγκριση με την πατρίδα σας, τη Γερμανία, εάν ήταν αναγκασμένη η Γερμανία να κάνει μειώσεις του ελλείμματος της τάξης του 6,5% του ΑΕΠ, τότε οι περικοπές θα αντιστοιχούσαν σε 100. 60 δισεκατομμύρια ευρώ. Το πρωτογενές έλλειμμα εδώ στην Ελλάδα μειώθηκε μέσα σε δύο χρόνια από 24 δισεκατομμύρια ευρώ σε 5 δισεκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή από 10,5 σε 2,5 το ακαθάριστο εγχώριο προϊόντος. Ο δημόσιος τομέας μειώθηκε δραστικά. Ο αριθμός των δημοσίων υπαλλήλων είναι κατά 200.000 μικρότερος σε σύγκριση με το 2009. Το εισόδημα των εργαζομένων και των συνταξιούχων έχει μειωθεί επίσης σε μεγάλο βαθμό. Παντού γίνονται περικοπές. Παντού κάνουμε περικοπές. Και εδώ στο Κοινοβούλιο. Κατά 50% μειώθηκαν τα λειτουργικά έξοδα της Βουλής των Ελλήνων, όπως και οι μειώσεις στη βουλευτική αποζημίωση αγγίζουν το 50% για τους Έλληνες βουλευτές. Αλλά πάνω απ' όλα οι προσπάθειες είναι, όπως είπα, του ελληνικού λαού που κάνει τεράστιες θυσίες. Και θέλω στο σημείο αυτό να υπογραμμίσω ότι οι Έλληνες, κύριε Πρόεδρε, εργάζονται σκληρά. Δεν σας κρύβω ότι οργιζόμαστε και οργίζομαι και εγώ όταν διαβάζουμε ή ακούμε ισχυρισμούς ορισμένες φορές αλλά κάποιες φορές και δηλώσεις πολιτικών ότι δήθεν οι Έλληνε δεν δουλεύουν αρκετά, ότι οι Έλληνες είναι τεμπέληδες. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΟΣΑ που δημοσιεύονται κάθε χρόνο οι Ιταλοί εργάζονται κατά μέσο όρο 1.778 ώρες ετησίως. Οι Πορτογάλοι εργάζονται 1.714 ώρες. Οι Ισπανοί εργάζονται 1.663 ώρες. Οι Γάλλοι εργάζονται 1.554 ώρες οι Γερμανοί εργάζονται 1.419 ώρες και οι Έλληνες, οι Έλληνες εργάζονται 2.109 ώρες. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΣΑ, μόνο οι Νότιο Κορεάτες εργάζονται περισσότερο από τους Έλληνες. Την αμέσως επόμενη θέση είναι οι Έλληνες σε ό,τι αφορά τις ώρες εργασίας ετησίως. Γι' αυτό λέω ότι ο ελληνικός λαός εργάζεται σκληρά. Εδώ στο Κοινοβούλιο πήραμε αυτά τα δύο χρόνια αποφάσεις δύσκολες και οδυνηρές. Και δεν σας κρύβω ότι πήραμε αποφάσεις που πολλές φορές έρχονται σε σύγκριση ακόμη και με αυτά που πιστεύουμε, με την ιδεολογία μας και τα πολιτικά μας πιστεύουμε. Πήραμε όμως και παίρνουμε τις αποφάσεις αυτές για να προφυλάξουμε πρώτα απ' όλα τη χώρα μας από την χρεοκοπία, για να την προφυλάξουμε από την ολική καταστροφή. Πήραμε τις αποφάσεις αυτές έχοντας ταυτόχρονα επίγνωση, και το υπογραμμίζω αυτό, επίγνωση των υποχρεώσεων και των δεσμεύσεών μας απέναντι στους εταίρους μας στην Ευρωζώνη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά. Θα πρέπει όμως πιστεύω να έχουν όλοι υπόψη ότι η Ελλάδα, ο ελληνικός λαός δικαιούται να έχει τον σεβασμό για την τεράστια προσπάθεια που καταβάλλεται εδώ, δικαιούται να έχει αυτόν από τους άλλους αυτόν τον σεβασμό για τις θυσίες τις οποίες υποβάλλεται. Και θα ήθελα να κλείσω με μια επισήμανση που αποτελεί πεποίθησή μου και είμαι σίγουρος ότι δεν είναι μόνο δική μου πεποίθηση. Η οικονομική κρίση στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες χώρες στην Ευρώπη δεν πρόκειται να ξεπεραστεί μόνο με δημοσιονομικά μέτρα, με περικοπές και μειώσει των ελλημάτων. Οι περικοπές οδηγούν σε βαθιά ύφεση και οδηγούν σε εκτείναξη της ανεργίας. Και εδώ αλλά και σε άλλες χώρες όπως η Πορτογαλία, η Ιρλανδία, η Ισπανία, η Ιταλία και όχι μόνο. Είναι αναγκαίο πιστεύω να δοθεί άμεσα ιδιαίτερο βάρος στην ανάπτυξη. Αυτό πρέπει να αντιληφθούν και όλες οι πολιτικές ηγεσίες στην Ευρώπη. Χρειαζόμαστε ανάπτυξη. Και μέχρι σήμερα εκτιμώ ότι οι ηγεσίες στην Ευρώπη συζητούν πολύ λίγο για την ανάπτυξη και πράττουν ακόμη λιγότερα για αυτήν. Είναι αδύρυτη ανάγκη όμως να υπάρξουν συγκεκριμένες αποφάσεις, προγράμματα, πρωτοβουλίες για να έχουμε την πολυπόθητη ανάπτυξη. Μόνον έτσι άλλωστε θα αντιμετωπιστεί και το τεράστιο πρόβλημα της ανεργίας και ιδιαίτερα της ανεργίας των νέων. Ανεργίας των νέων που δυναμητίζει τα θεμέλια της κοινωνικής συνοχής και θέτει σε κίνδυνο το ίδιο το όραμα της ΕΕ. Ευρώπης. Μόνον έτσι θα υπάρξει βάσιμη ελπίδα για το μέλλον. Κύριε Πρόεδρε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον περιμένουμε, αναμένουμε απόψε την δική σας ομιλία. Σας καλώ λοιπόν στο βήμα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητές κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι, χαίρομαι που μπορώ σήμερα να σας μιλήσω ως πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά και ως χαμανός ευρωβουλευτής.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 Ε, πρέπει να σας πω ότι αν κοιτάξω εδώ ποιοι είναι μπροστά μου, έχω την εντύπωση ότι σε τελική ανάμεστη είμαστε παλιοί ευρωβουλευτές όλοι μεταξύ μας οι οποίοι καθόμαστε εδώ και είμαστε έτοιμοι να μιλήσουμε. Ε, ε χαίρομαι ιδιαίτερα να πω και, και πάρα όλα χαίρομαι που βλέπω τόσους συναδέλφους, παλιούς συναδέλφους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, φίλους όλους, τους οποίους μπορώ σήμερα να δω εδώ και να συγχαρώ και να μιλήσω μαζί τους. Με πονάει. Με πονάει που πρέπει να δω ότι ένα κράτος το οποίο μια στιγμή ήταν υπέρ της Ευρώπης αυτή τη στιγμή είναι απογοητευμένο και είναι εκνευρισμένο, είναι μέσα στο θυμό και στρέφει τα νότα του στην Ευρώπη. Οι εικόνες από ανθρώπους οι οποίοι καίνε τις ε, σημαίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους δρόμους της Αθήνας. Αυτά ήταν εικόνες τις οποίες πραγματικά είδα και αισθάνθηκα ότι έχω τροφή προσωπικά ότι η ευρωπαϊκή σημαία η οποία είναι μια σημαία ένα σύμβολο της ειρήνης και της ενότητας της δημοκρατίας, της αλληλεγγύης ότι αυτή ακριβώς αυτή η σημαία για ορισμένους μέσα στην πατρίδα σας και όχι μόνο εδώ αλλά και σε άλλα κράτη της Ευρώπης ξαφνικά είναι το σύμβολο για το γεγονός ότι υπάρχει εγωισμός και είναι απόψεις οι οποίες εναρνητικές θα πρέπει να ανοίξει τα μάτια όλων μας για τη δραματική κατάσταση ισχύει στην Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη πιστεύω. Με πονάει προσωπικά ότι πρέπει να δω ότι όλα αυτά τα χρόνια, τα, οι δεκαετίες καλής επαφής μεταξύ Ελλάδο και Γερμανία, μέσω αυτή τη κρίση, αλλά αργά αλλά σταθερά φαρμακώνονται οι σχέσεις Οι σχέσει μα. Οι σχέσεις ε, ε, των δύο εθνών και κρατών δεν ήταν ποτέ εύκολο. Πρέπει να πω ότι η, αν θέλετε, η ζωή του κυρίου Παπούλια, που πούμε, του Προέδρου της Δημοκρατίας, είναι ένα παράδειγμα των σχέσεων των δύο κρατών. Er Ήταν 14 ετών όταν για πρώτη φορά στην Ήπειρο όπου ζούσε, ε, είπε ότι θα έπρεπε να βοηθήσει τον ελληνικό um απελευθερωτικό στρατό ε, για να αντιμετωπίσει τους Γερμανούς κατακτητές ε, η Γερμανία του Χίτλερ είχε καταλάβει την Ελλάδα, υπήρχαν τραγικές εξελίξεις προκειμένου και γεγονότα. Αργότερα, κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1960, ο κύριος Παπούλιας μπόρεσε να βρει το δρόμο στη Γερμανία και να σπουδάσει νομικά από τον αντιστασιακό αν θέλετε εκείνη τη εποχή έγινε ένας φίλος ένας φίλος της δικής μου της πατρίδας και νομίζω ότι αυτό σημαίνει ότι ο δικός σας ο πρόεδρος της, κοινοβου... Ε, Δημοκρατίας είναι ένας από εκείνους ο οποίος συγχώρησε τα παράδεκτα τα οποία είχαν συμβεί κατά την περίοδο της κατοχής και έδωσε το χέρι για ένα χέρι βοηθείας και αλληλεγγύης. Εγώ προσωπικά πρέπει να σας πω ότι στην Ελλάδα έχω πάρα πολλούς φίλους σε αυτή την θαυμάσια χώρα και πρέπει να σας πω ότι είναι μια ανάγκη καρδιάς να επουλώσουμε τα τραύματα, να μπορέσουμε πραγματικά να μιλήσουμε εδώ και τώρα ε, για πραγματικές ε, αλήθειες και να μην μιλάμε με γενικότητες, να έχουμε διάλογο, συνεργασία και να μην έχουμε όλα αυτά τα κλισέ τα οποία πιστεύουμε ότι χαρακτηρίζουν τις σχέσεις και τους λαούς μας. Θέλω να λείπω στην Ευρώπη, θα γίνουμε εταίροι και όχι αντίπαλοι. Μερικές φορές έχω την εντύπωση ότι είναι περισσότερο και ένα είδος του τόνου, δηλαδή είναι ένας κακός στυλ και πολύ περισσότερο περιεχόμενο αυτό το οποίο δει. Να σας πω κάτι, αδιαφόρος του πόσο επιθετική ρητορία μπορεί να χρησιμοποιεί κανείς και αδιαφόρος ε, όλων εκείνων οι οποίοι σηκώνουν το δάχτυλο και προσπαθούν να δώσουν συμβουλές και η Γερμανία πάντοτε ήταν αλληλέγγυα. Αυτό μην το ξεχνάμε. Το Γερμανικό Κοινοβούλιο χθε ε, συμφώνησε για το δεύτερο πακέτο βοήθειας με 419 ψήφους, 490 ψήφους, συγγνώμη. Η Ομοσπονδική Δημοκρατία της Γερμανίας εγγυάται αυτή τον, τον σταθεροποιητικό μηχανισμό με, από, τα οποία, από τα 800 εκατομμύρια που χρειάζεται τα 211. Είναι περισσότερο από τον προϋπολογισμό της ε, Γερμανίας της ίδιας. Ένα όμως είναι σαφές. Ουδέποτε, ουδέποτε πρέπει η βοήθεια του ενός ε, να καταστρατηγεί το σεβασμό, την τιμή και την αξιοπιστία του άλλου. Γι' αυτό το λόγο ακριβώς θα ήθελα να ελπίζω ότι θα είμαστε εταίροι στις προσπάθειές μας και στο διάλογο τον οποίο θέλουμε να αναπτύξουμε. Ίσως, ε, έχουμε την εντύπωση ότι είναι ένα γερμανοελληνικό πρόβλημα. Είναι περισσότερο από αυτό. Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης πολύ συχνά, um πάρα πολύ συχνά, εδίστασαν να πάρουν την σωστή απόφαση την κατάλληλη στιγμή. Λόγω αυτής του δισταγμού, της αβελτηρίας, στην Ευρώπη ε, δημιουργήθηκε μια ατμόσφαιρα η οποία καταρχάς έδωσε τη δυνατότητα να αρχίσουν αυτοί οι εθνικιστικοί εγωισμοί και όλες αυτές οι ατασταλίες και οι τραγικές πράξεις. Ο Μάριο Μόντι πριν από λίγες μέρες είπε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο των Μασίνες και έκρουσε τον κόδωνα του κονδύνου και είπε τα στερεότυπα, οι προκαταλήψεις οι οποίες υπάρχουν, οι τα εικόνε των εχθρών, όχι μόνο μεταξύ Ελλήνων και Γερμανών, αλλά όλοι σε όλη την Ευρώπη έχουν και παίζουν τον πρώτο ρόλο. Κυρίε και κύριοι, όλοι εσεί, οι οποίοι είστε συνάδελφοι σε αυτό το κοινοβούλιο, εμά που είμαστε συνάδελφοι στα Εθνικά Κοινοβούλια και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, παρακαλώ όλου εμά να μην ξαναπέσουμε μέσα στα παλιά κλισέ και στι παλιέ προκαταλήψει, στου εθνικισμού κατά του ενό, του ενό κατά του άλλου. Ο Κυρίες και κύριοι, μόνο ένα κάθε φορά έφερε και επέφερε. Ατυχία. Ατυχία για όλους τους λαούς στην Ευρώπη. Πόνο και δυστυχία. Αγαπητοί συνάδελφοι, σήμερα είμαι εδώ στην Αθήνα γιατί σε εσά τους εκπροσώπους του ελληνικού λαού και ταυτόχρονα και στο ελληνικό ε, λαό να πω πόσο το σέβομαι ξέρω um ε, τις δυσκολίες, το um άχθος το οποίο πρέπει να σηκώσετε, ε, τις δύσκολες αποφάσεις, τις τραυματικές αποφάσεις τις οποίες πήρατε όλους αυτούς τους μήνες και θα πάρετε και σήμερα το βράδυ. Ο συνάδελφο καταλαβαίνω πόσο δύσκολο είναι για όλους εμάς τους πολιτικούς, για μένα, για σας, να πάρουμε αποφάσεις οι οποίες όταν έχουμε, ε, ε, οι οποίες ξεπερνούν τον ορίζοντα μέσα στον οποίο θα μπορεί κανείς να εκλεγεί. Ξέρω ότι πρέπει να πάρει πάρετε αποφάσεις οι οποίες πιθανόν, πιθανόν να σας κοστίσουν την έδρα σας στο Κοινοβούλιο. Η κατάστασή σας είναι παρόμοια ε, με πολλούς άλλους βουλευτές σε όλα τα άλλα κοινοβούλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν και εκπρόσωποι σε άλλα κοινοβούλια, τα οποία αυτή τη στιγμή, τη στιγμή που υπερψηφίζουν τη βοήθεια στην Ελλάδα, παίζουν την έδρα τους και τη δυνατότητα επανεκλογής τους. Παρόλα αυτό όμως, παρόλα αυτή τους ενδιασμούς, το πρόβλημα, πήρανε αυτή τη δύσκολη απόφαση και ε, κινήθηκαν προς τη σωστή κατεύθυνση. Πήρατε δύσκολες αποφάσεις εσείς και αναλάβατε και αντίστοιχες ευθύνες. Νομίζω ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό παίξατε έναν πατριωτικό ρόλο. Αλλά έχω και μεγάλη κατανόηση για όλους εκείνους που είναι στους δρόμους και συνεχώς κινούνται κατά και, και κατανοώ και όλους εκείνους οι οποίοι είναι έξαλλοι επειδή τους κόψανε δηλαδή ε, τους μισθούς. Για συνταξιούχους οι οποίοι πλήρωναν για τη σύνταξή τους και ξαφνικά τους μειούται αυτοί. Καταλαβαίνω τους νέους ανθρώπους οι οποίοι φοβούνται για το μέλλον τους και ενώ τους είχε εξαπατήσει κανείς. Και να πω κάτι για την ενεργία των νέων. Το γεγονό ότι η μοντέρνα οικονομία της Ευρώπης το επιτρέπει ότι ένα 40% των νέων ανδρών και γυναικών δεν έχουν δουλειά δεν είναι μόνο ντρομή, είναι αυτό το οποίο καταστρατηγεί τη δημοκρατία σε όλη την Ευρώπη. Πώ θα μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να αποκτήσουν εμπιστοσύνη σε αυτή την κοινωνική μας δομή αν δεν του δίνουμε αυτή τη στιγμή μέλλον. Αυτό δεν είναι ελληνικό πρόβλημα, είναι ευρωπαϊκό πρόβλημα. Η καταπολόμηση ανεργία των νέων είναι μια πρόκληση για όλου. και περιμένω αν ο κύριο Παπαδήμο αύριο έρθει στην Βρυξέλλες ότι με την Κομισιόν, με του αρμόδιους επιτρόπους να μπορέσει να μιλήσει και να συζητήσει και να πει ότι τα μη χρησιμοποιηθέντα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να χρησιμοποιηθούν για την, ε, να εξευρεθούν θέσεις εργασίας και στην Ελλάδα και σε όλα τα άλλα κράτη Ευρώπη, θέσει εργασία για Δεν έχω όμω κατανόηση κύριε και κύριοι για όλου εκείνου που δεν πληρώνουν φόρου. Και δεν έχω καμία κατανόηση για όλου εκείνου οι οποίοι παράνομα όλα τα χρήματά του τα βγάζουν εκτό ε, Ελλάδος. Ζητώ από τους πλούσιου οι υπάρχουν στην Ελλάδα. Δώστε στην πατρίδα σας κάτι πίσω από όλα αυτά το οποίο η πατρίδα σας σας έδωσε. Είναι η πατριωτική σας ευθύνη και υποχρέωση. Απαιτείται μια εσωτερική συνοχή σε ένα λαό. Απαιτείται πραγματικό να έχουμε μια πολιτική κουλτούρα η οποία από μέσα να δομεί και να δομείται για να ξεπεράσει κανείς και την κρίση και να επιδείξει αλληλεγγύη και να ζητήσει αλληλεγγύη από την Ευρώπη. Κυρίες και κύριοι, επιτρέψτε μου για αυτό το λόγο να κάνω κάποια σχόλια σε σχέση με θέματα τα οποία για εγώ είμαι απόλυτα επιπλέον για την ορθότητά του. Η Ελλάδα πρέπει να μείνει στο ευρώ. Αυτό είναι το καλύτερο για το συμφέρον της δικής σας, της πατρίδας και της Ευρώπης. Αυτή τη στιγμή είμαστε όλοι στο ίδιο πλοίο, μέσα. Μόνο μαζί μπορούμε πραγματικά να ξεπεράσουμε τη φορτούνα και την τρικυμία. Η Ευρώπη είναι το κοινό μας μέλλον. Um πρέπει να κάνουμε το παν για να μπορέσουμε να μείνουμε και να μην επιτρέψουμε να καταστρεφεί ή να καταστραφεί το ευρώ. Αν σώσουμε το ευρώ, δεν είναι θέμα ποιο θα είναι το υφή του ευρώ με την οποία πληρώνουμε, αν είναι νόμισμα ή χαρτί, ούτε αν πάμε ε, τώρα αυτή τη στιγμή για διακοπές θα πρέπει να πάμε να αλλάξουμε και να αποκτήσουμε συνάλλαγμα. Είναι ότι αν αποτύχει αυτό το κοινό μας νόμισο η Ευρώπη με ένα δραματικό τρόπο πραγματικά από οικονομικής και πολιτικής πλευράς θα χάσει στα πλαίσια του διεθνούς ανταγωνισμού μέσα στον οποίο βρισκόμαστε και πρέπει να επιβιώσουμε μέσα σε αυτόν. Όλοι εμείς πρέπει να καταλάβουμε ότι μόνο αν είμαστε μια ισχυρή, ένα ισχυρό κομμάτι του κόσμου ολόκληρος, αν κινηθούμε όλοι μαζί, ε, μπορούμε κάτι να κάνουμε. Αν κατακαιρματιστούμε θα γίνουμε αδιάφοροι, μικροί και περιθωριακοί. Σώζουμε το ευρώ για να είμαστε σίγουροι να ε, προχωρήσουμε στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Εγώ πιστεύω ότι είναι το πιο ενδιαφέρον project της εποχής μας. Αν θα μπορέσουμε πραγματικά να έχουμε μια ευρώ. Ευρώπη με συνοχή. Σώζοντας το ευρώ, ταυτόχρονα το είναι αν θα σώσουμε και την ευρωπαϊκή ιδέα και το ιδεώδες. Το ευρωπαϊκό ιδεώδες είναι αντιμετωπίζω προβλήματα και προκλήσεις με το διάλογο και με τη συνένεση. Δεν επιτρέπω το δίκαιο του ισχυρότερου, αλλά το δίκαιο του ισχυρότερου είναι το ισχυρό του δικαίου. Αυτό σημαίνει η δημοκρατία. Αυτό θα πρέπει να είναι η βάση του τρόπου με τον οποίο κινούμαστε. Τώρα, αν είμαστε διατεθειμένοι πραγματικά να βάλουμε το κοινό καλό πάνω από το μεμονωμένο, του μικρού κράτους υπεράνω, του κομματικού πάνω από το κοινό, για να μπορέσω πραγματικά να βοηθήσω το σύνολο και όχι το επιμέρους. Επιτρέψτε μου να πω επίσης ότι αν κάνουμε μια πολιτική η οποία είναι καθαρά πολιτική εξοικονόμησης, ε, ε, ναι, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, αλλά δεν πρέπει έπρεπε αυτή τη στιγμή να ξεχνάμε ότι το χρέο θα πρέπει να ελεγχθεί. Αλλά το χρέο είναι και κάτι το οποίο θα πρίνει και μια δικαιοσύνη και για τι μελλοντικέ γενιέ. Δεν μπορούμε να του αφήσουμε χρέη επί Αλλά εδώ και τώρα η συζήτηση ασχολείται μόνο για την επιβολή και για τα πακέτα διάσωση και εξοικονόμηση. Αυτό σημαίνει ότι η ανάπτυξη είναι ένα παράγοντας ο οποίο σε πάρα πολλά κράτη και ιδιαίτερα στην Ελλάδα πρέπει να το πω, κοντεύουμε να την πνίξουμε την ανάπτυξη. Η οικονομία έχει πάψει να κινείται, έχει πάψει να υπάρχει. Αν αυτή τη στιγμή έχουμε μία ύφεση, πώς θα μπορέσουμε μέσα από μία ύφεση τέτοιου είδους κράτη να τα βοηθήσουμε να εξαλείψουν τα χρέος τους. Η Ελλάδα έχει πληρώσει πολύ. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Πρέπει το Ευρωπαϊκό Κοινόλιο από την αρχή αυτής της κρίσης και το έχει πει ότι θα πρέπει να κάνουμε ότι θα πρέπει ναι να περιοριστεί το χρέος αλλά ταυτόχρονα συνδυαστεί με ανάπτυξη και αναπτυξιακά μέτρα. Για τους περισσότερους βουλευτές, κυρίες και κύριοι, λένε ότι ο ισοσκελισμένος προϋπολογισμός δεν θα πρέπει να είναι εις βάρος της κοινωνικής δικαιοσύνης. Πρέπει να υπάρχει αυτό που λέμε φέρνες. Δεν μπορεί οι πιο ασθενείς πραγματικά να σηκώσουν το άχθος, το βάρος της κρίσης. Η οικονομική κρίση οδήγησε στη φτώχεια, στην ένδια και στην κρίση. Αλλά αν συνεχίσουμε να σφίγγουμε αυτή τη στρόφικα συνεχώς, η κατάσταση θα έχει Η Ευρώπη δεν είναι, αν θέλετε, είναι μια κοινωνία της αλληλεγγύη, Δεν είναι μια κοινωνία με στην οποία ύψιστο αγαθό είναι το εξοικονομή χρήματα. Πρέπει πραγματικά να δούμε και η Ελλάδα χρειάζεται ενάψματα για ανάπτυξη. Πρέπει η Ελλάδα αυτή τη στιγμή να βρει εργασίε, jobs λέει ο Jobs οι οποίοι πραγματικά να σημαίνουν ότι θα δημιουργηθεί κίνηση μέσα στη χώρα, θα μπορέσει να υπάρχει αγορά, θα πρέπει να είναι αυτή τη στιγμή ανάπτυξη και ανάγκη. Οι άνθρωποι εδώ πέρα και η, οικονομία σε αυτή τη χώρα χρειάζεται μια προοπτική. Και επιτρέψτε μου να σα πω, ε, να σα κάνω κάποιε μικρέ προτάσει από τη δική μου την οπτική. Σα είπα, είπα προηγουμένω, μέσα στα πλαίσια του Κοινωνικού Ταμείου και του Ταμείου Αλληλεγγύης θα πρέπει να κινητοποιηθούν για την Ελλάδα, για να βοηθήσουμε θέσει εργασίε μέσω επενδύσεων στι υποδομέ. Ταυτόχρονα, μικρομεσαίε επιχειρήσει χρειάζονται και αποκτούν δάνεια. Και γι' αυτό το λέω χαίρομαι που η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θέλει να αναπτύξει ένα πρόγραμμα μικροδανείων για την Ελλάδα. Πρέπει να βοηθήσουμε σε ανθρώπου, μικρομεσαίου οι οποίοι θέλουν να επενδύσουν πρέπει να βοηθηθούν. Δεν θα πρέπει να περιμένουν τα δάνεια. Τα δάνεια θα πρέπει σχεδόν να του προσφερθούν για να ξαναμπούν μέσα στην αγορά και να δημιουργήσουν ζήτηση. Και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να έχουμε μια διοίκηση η οποία να λειτουργεί ευρύθμω. Και οι ανακατατάξει οι οποίε θα πρέπει να γίνουν, αυτό το ξέρετε καλύτερα από μένα, πρέπει να γίνουν. Χαίρομαι ιδιαίτερα που η Κομισιόν το κατάλαβε. Χθε μίλησα με τον κύριο Μπαρόζο και μίλησα διαμακρών και θέλω να ελπίζω ότι τα μέτρα τα οποία θα πάρει η Task Force όταν θα έρθει στην Ελλάδα να βοηθήσει ακριβώς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να τους υποστηρίξει. Και πάνω απ' όλα να βοηθήσει και το δημόσιο τομέα στην ανακατάταξη και αναδιάρθρωση. Υπάρχουν υπάρχουν ευρωπαϊκά χρήματα. Τα ευρωπαϊκά χρήματα όμως δεν μπορούμε να τα βάλουμε σε διάφορα ταμεία, πρέπει να τα επενδύσουμε και η επένδυση αυτού του χρήματος πρέπει να γίνει με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο. Εάν έχουμε ε, γραφειοκρατικά εμπόδια τα οποία απεμπολίσουμε, τότε χωρίς αμφιβολία οι επενδύσεις δεν θα φτάσουν μόνο στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά θα έχουμε και τους μεγάλους επενδυτές οι οποίοι θα έρθουν. Οι μεγάλοι επενδυτές θα μπορούσαν να μπουν ας πούμε στην ηλιακή ενέργεια. Είναι το ιδανικότερο μέρος αν θέλετε πραγματικά να επενδύσει κανείς σε μια νέα τεχνολογία και μια νέα βιομηχανία η οποία απαιτείται και χρειάζεται η ηλιακή ενέργεια.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 το πρόγραμμα Ήλιος, το οποίο είχε αρχίσει να λειτουργεί στα πρόγραμμα του προγράμματος 2020 για να δημιουργήσει πράσινες θέσεις εργασίας, δεν πρέπει να μείνει μόνο στα χαρτιά της Ευρώπης του 2020. Πρέπει επιτέλους να αρχίσει να λειτουργεί και να χρησιμοποιείται, να δώσει επενδύσεις και να δημιουργήσει θέσεις εργασίας. Και θέλω να πρεστήσω, για να χρηματοδοτηθεί αυτό, είμαι πραγματικά υπέ να έχουμε project bonds, τα οποία να δημιουργηθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση χαίρομαι που η Κομισιόν αποφάσισε την Πέμπτη να δώσει και να συζητήσει τέτοιου είδου projects μέσα στα πλαίσια του Συμβουλίου Κορυφή. Επιτέλου να σα πω κάτι. Ένα πρόγραμμα για το οποίο πιστεύω εγώ είναι η Ένωση για, την, ε, για τη Μεσόγειο. Στη Νότια Αφρική εκατοντάδε χιλιάδε άνθρωποι θέλουν να δημιουργήσουν ένα νέο μέλλον. Ο πραγματικό εταίρο είναι τη Βορείου Αφρική είναι η Νότιο Ευρώπη. Και τι χρειάζονται οι άνθρωποι στη Βόρειο Αφρική πάνω απ' όλα. Χρειάζονται επενδύσεις στις υποδομές, ε, στα νοσοκομεία, στα σχολεία, στα πανεπιστήμια, σε μια πραγματική αγροτική παραγωγή η οποία να έχει μέλλον και βάθος. Ποιο μπορεί να τους βοηθήσει, ποιο μπορεί να είναι εκείνος ο οποίο θα δώσει την τεχνορωσία, το know-how, μα ο νότος της Ευρώπης. Όχι μόνο η Ευρώπη. Δεν είναι μόνο από πλευρά πολιτική, αλλά και από γεωγραφική πλευρά. Είναι ένα πλεονέκτημα να είναι εκεί, εκεί που είναι ε, και αν πραγματικά έχουμε μια ένωση των μεσογειακών κρατών θα μπορέσουμε να κάνουμε κάτι και να είναι το μέλλον του 21ου αιώνα. Γιατί? Γιατί αυτό είναι κάτι και ρωτώ γιατί δεν κάνουμε κάτι παραπάνω προς αυτή την κατεύθυνση με μεγαλύτερο κέφι και ενέργεια η Ελλάδα έχει δυνατότητε. Οι δυνατότητες όμως αυτές κύριε και κύριοι είναι δυνατότητε οι οποίε πρέπει κάποτε να χρησιμοποιηθούν. Και πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και επαναλαμβάνω ε, δεν πιστεύω ότι είμαι εδώ πέρα να στέλνω μόνο έναν πρέσβο που να πει εξοικονομείτε, εξοικονομείτε, εξοικονομήστε. Πρέπει το μήνυμα να είναι έχει νόημα να γίνουν επενδύσει, όχι μόνο για του Έλληνε, αλλά και για ξένου. Και αν η Ελλάδα τα πάει καλά και είναι καλά τότε θα είναι και άλλοι Ευρωπαίοι οι οποίοι θα έχουν ένα ενδιαφέρον να επενδύσουν στην Ευρώπη. Εδώ και τώρα υπάρχουν πολλές συζητήσεις για την κρίση αυτής της Ευρώπης και του ευρώ. Δεν νομίζω ε, όμως ότι αυτό ισχύει. Το ευρώ, όπως ε, βλέπετε, έχει μια σταθερή αξία προς τα έξω, τη συναλλαγματική αξία. Γιατί, διότι από τη μία μεριά έχουμε μια κρίση επικρίσεως την οποία συζητάμε, αλλά έχουμε ένα νόμισμα του εξακολουθεί να έχει μια σταθερή εξωτερική αξία. Γιατί, Γιατί οι Ηνωμένε Πολιτείε της έχουν με, μεγαλύτερη υπερχρέωση από ό,τι εμείς ε, και ίσως και ένα πιο περιορισμένη οικονομική ανάπτυξη ανάπτυξη από εμά, αλλά οι επενδυτέ που πάνε στην Αμερική, στι Ηνωμένε Πολιτείες δηλαδή και όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωζώνη. Νομίζω ότι δεν θα πρέπει να έχουμε αυτά πάτε εν προκειμένου. Οι Ηνωμένε πολιτείε τη Αμερική έχουν σε αντίθεση με την Ευρωζώνη, δεν έχουν να κάνουν και να αντιμετωπίσουν με το γεγονό ότι υπάρχει περίπτωση αυτό το νόημα να καταστραφεί ή να μην υπάρξει. Μην έχουμε αυτά πάτες. Οι οικονομικές αγορές είναι κάτι το οποίες παίζουν με το τέλος του ευρώ και θα βγάλουν χρήματα. Άρα το μόνο το οποίο μπορούμε να κάνουμε προκειμένου είναι να υπεραμεινθούμε του ευρώ. Και με αυτόν τον τρόπο, αν υπεραμεινθούμε του ευρώ, πρέπει να κάνουμε και αυτό το ξέρουμε και είναι η δυνατότητα να πούμε επισήμως αφήστε το, δεν έχει νόημα. Η Ευρωζώνη εδώ είναι και θα μείνει αλληλέγγυα και θα παραμείνει έτσι όπως είναι. Αυτό είναι το μήνυμα το οποίο εγώ για άλλη μια φορά θα πω την Πέμπτη στη Σύνοδο Κρατών ε, και ε, Κυβερνήσεων. Και θέλω να ελπίζω ότι και εσείς μαζί με μένα θα έχουμε μεγαλύτερη διευθέτηση των αγορών γιατί η χρηματοπιστωτικές αγορές θα πρέπει να το έχουμε και αυτό σημαίνει θα πρέπει να έχουμε και μια φορολόγηση ε, των ανταλλαγών και συναλλαγών στα χρηματιστήρια. Δεν είναι δυνατόν κυρίες και κύριοι όλοι εκείνοι οι οποίοι μέσα από τη σπέκουλα, μεγάλες τράπεζες, μεγάλες ασφαλιστικέ εταιρείε, τα μεγάλα hedge funds, ε, ε, από το 2008 και μετά έχουν βγάλει πάρα πολλά λεφτά. Δεν είναι δυνατόν ε, ότι αυτοί οι οποίοι, οι μεγάλοι επενδυτικοί οίκοι, τα μεγάλα Ινστιτούτα επενδύσεως, ε, να μην συμμετάσχουν πραγματικά στις επιπτώσεις οι οποίες υπάρχουν. Γι' αυτό ζητώ και απαιτώ για άλλη μια φορά και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το έκανε με ένα πολύ ουσιαστικό τρόπο και το παρουσίασε και η συνάδελφος κυρία Ποδηματά. Πρέπει πραγματικά να έχουμε μια φορολόγηση των χρηματοπιστωτικών αλλαγών. Και αυτό να γίνει τώρα και όχι του Αγίου ποτέ. Κυρίες και κύριοι, αν έχουμε μια οικονομική ένωση, η οποία είναι και μια φορολογική ένωση και μια ένωση οικονομική και χρηματοπιστωτική, χρειάζεται ένα περισσότερο, ένα συν μέσα στο κοινοβούλιο. Τα τελευταία λεφτά άκουσα, θα το μάθετε κι εσείς, ότι στην Ιρλανδία θα υπάρξει όσον αφορά την ε, φορολογική ένωση στην Ιρλανδία. Ο, ο, ο λαός της Ιρλανδίας θα ψηφίσει εν προκειμένου. Θα υπάρξει ένα δημοψήφισμα. Αλλά στην Ελλάδα ε, χρειαζόμαστε στο ευρωπαϊκό επίπεδο καθαρά, σε όλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για όλα τα μέτρα τα οποία παίρνονται στα πλαίσια αυτής της απόφασης, μια κοινοβουλευτική αξιοπιστία και επικύρωση. Όλα αυτά τα μέτρα πρέπει να επικυρωθούν και να μπουν και να γίνουν εθνικό δίκαιο, άρα θα περάσουν από τα εθνικά κοινοβούλια. Αν όμω ε, το Eurogroup, το, η Σύνοδος Κορυφής, κάθε φορά κάνει τέτοια μέτρα, τότε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει πραγματικά να έχει την νομιμοποίηση, να εισηγηθεί και να αποδεχθεί. Γι' αυτό το λόγο κυρίε και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι του Ελληνικού Κοινοβουλίου, πρέπει να καταλάβετε, δεν είμαστε αν θέλετε αντίπαλοι όσον αφορά τον κοινοβουλευτισμό στην Ευρώπη. Είμαστε εταίροι. Πρέπει τα 28 κοινοβούλια πραγματικά να πιστούν και να υπερψηφίσουν και οι Κομισιόν και 27 κυβερνήσει. Θα πρέπει να υπάρχει το εθνικό κοινοβουλευτισμό. Ναι, και εσεί είστε υπεύθυνοι για μια σειρά από πράγματα, αλλά όταν η κυβέρνησή σα, ω μέλο ε, των ευρωπαϊκών θεσμών, τότε εμεί ω Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είμαστε υπεύθυνοι για το ότι γίνεται ή όχι. Και αυτό είναι ένα αίτημα προ εσά. Επιτρέψτε μα μέσα ω πλαίσιο του κοινοβουλευτισμού να συνεργαζόμαστε και όχι να είμαστε αντιτιθέμενε ομάδε. Αγαπητοί συνάδελφοι, έχετε στη στιγμή που πρέπει πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά. Οι αποφάσει των τελευταίων ημερών, αν θέλετε, έβαλα τα χαρτιά πάνω στο τραπέζι πια. Εσείς δεχθήκατε και uh, υποψηφίσατε για πράξεις όπου περιμένουμε όλοι ότι θα τις υλοποιήσετε και θα τις στηρίσατε. Και όσο και αν είναι δυσάρεστα αυτά τα πράγματα, είναι κάτι το οποίο είναι ίδιο ενδιαφέρον και για σας. Ζητώ από όλου εσά, κύριε και κύριοι και ξέρω ότι είναι δύσκολο και ξέρω ότι σήμερα το βράδυ πρέπει πάλι να ψηφίσετε κάτι πολύ δύσκολο. Το πρόγραμμα αυτό αναδιαρθρώσεως θα πρέπει να το υπερψηφίσετε. Να αισθάνεστε προσεκτικά δεσμευμένοι προκειμένου, αδιαφόρο των επικειμένων εκλογών. Και πάνω απ' όλα να ξέρετε ότι και η νέα κυβέρνηση μετά από τι επόμενε εκλογέ θα πρέπει να είστε σίγουροι θα ακολουθήσει αυτό τον δρόμο των αλλαγών, των ακατατάξεων και των καινοτόμων ιδεών. Μόνο έτσι θα κερδίσει τα αξιοπιστία και εμπιστοσύνη. Αλλά κυρίε και κύριοι, σα δώσαμε και, διαβεβλε... και διαβεβαιώσει. Διαβεβαιώσει από τι οποίε μπορείτε να περιμένετε ότι θα εκπληρωθούν. Και πρέπει να σα πω και στο σημείο αυτό, και εγώ με το στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα είμαι σίγουρο ότι θα προσπαθήσω να τηρηθούν όλε οι υποχρεώσει και υποσχέσει έναντι τη Ελλάδο. Οποιοδήποτε μέτρο εκτό ή παραπλεύρο θα δημιουργήσει δημιουργήσει πρόβλημα σε όλους τους πολίτες. Οι πολίτες της Ελλάδος έχουν κάνει θυσίες. Αν αυτό το οποίο φτάσαμε τώρα και το κερδίσαμε, αν αρχίσουμε να το αμφισβητούμε, τότε αυτοί οι άνθρωποι για άλλη μια φορά θα αρχίσουν να αναρωτιούνται γιατί. Και όχι μόνο αυτό, αλλά θα πιστεύουν ότι οι θυσίες τις οποίες κάνατε ήταν και δεν θα είχαν νόημα. Πάνω απ' όλο όμως θα αρχίσουν να αμφισβητούν την έννοια της αλληλεγγύης της οποίας τους έχει επιδειχθεί από τους άλλους. Αυτό αν όλοι εμείς δεν τηρήσουμε όλοι τις υποχρεώσεις που έχουμε δώσει. Πιστεύω για το μεγαλύτερο και μιλώ για το μεγαλύτερο κεφάλαιο το οποίο διαθέτουμε κυρίες και κύριοι. Το μεγαλύτερο κεφάλαιο το οποίο δεν προσμετράται από πλευράς κεφαλαίου. Το μεγαλύτερο κεφάλαιο είναι η εμπιστοσύνη. Εμείς σας εμπιστευόμαστε. Αλλά εσείς πρέπει να εμπιστεύεστε εμάς. Αν αυτή η αμοιβαία εμπιστοσύνη οδηγεί στο να κινητοποιηθούμε, τότε θα μπορέσουμε να κερδίσουμε και την εμπιστοσύνη των ανθρώπων. Και τότε θα έχουμε και την εμπιστοσύνη των ανθρώπων και θα το κερδίσουμε αυτή την εμπιστοσύνη, εάν πραγματικά τους δώσουμε μία ελπίδα, μία προοπτική ελπίδος. Η Ελλάδα δεν είναι μόνη της. Τα άλλα κράτη της Ευρώπης στέκονται πίσω από την Ελλάδα. Η Ελλάδα πρέπει να ξέρει ότι ναι, πρέπει να περάσει πολύ σκληρά και αυστηρά μέτρα και να τα αποδεχθεί. Πρέπει δύσκολα και μέτρα τα οποία πονάνε να τα αποδεχθεί και να ακολουθήσει αυτό τον ακαθόδη δρόμο. Αλλά σας λέω ότι πρέπει να ξέρετε και αυτό το το εκπροσωπώ εγώ σε Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εσείς οι Έλληνε, δεν είστε μόνοι. Είμαστε στο πλευρό σα, γιατί πιστεύουμε στις δυνατότητες αυτού του κράτους και αυτής της χώρας. Το μεγάλο και υπερήφανο έθνο σα, κύριε και κύριοι ξεπέρασε τους Ναζί. Το υπερήφανο αυτό κράτος μπόρεσε να ξεπεράσει τον εμφύλιο που ακολούθησε. Το υπερήφανο κράτος, το έθνος, η χώρα σας, το 1974 μπόρεσε να ξεπεράσει μια δικτατορία και να μπει πάλι στον εκδημοκρατισμό του Νότου της Ευρώπης. Η χώρα σας δεν είναι μόνο η χώρα η οποία στο παρελθόν στους αρχαίους χρόνους δημιούργησε τη δημοκρατία και στον 20ο αιώνα έκανε πάρα πολλά για τη δημοκρατία στην Ευρώπη μέσα. Για αυτή τη συνεισφορά εσείς η Ευρώπη είναι υποχρεωμένη να σας είναι πάντοτε ευγνώμων και είναι. Αλλά μέσα σε αυτό το πλαίσιο οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να πιστέψουν στην ευρωπαϊκή προπτική της χώρας Στο μέλλον της Ελλάδος και να αυτό να το, αυτού να υπεραμεινθούν. Εγώ πιστεύω, το πιστεύω αυτό. Είμαι πεπισμένο ότι αυτή η χώρα, εάν είμαστε όλοι μαζί, με εσείς ως λαός και, ε- και εσείς με όλους εμάς, με όλους τους λαούς της Ευρώπης μαζί, είμαι πεπισμένος ότι τότε η Ελλάδα πραγματικά έχει ένα μεγάλο, ένα λαμπρό μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον ε, κύριο Μάρτιν Σόλτς και υπογραμμίζω την αισιοδοξία του. Πρέπει να πιστεύουμε πράγματι στις δυνατότητες και πιστεύουμε κύριε Σούλτς εδώ στις δυνατότητες αυτού του λαού. Θα ακολουθήσουν τώρα σύντομε τοποθετήσεις τριών λεπτών από την δεύτερη αντιπρόεδρο της Βουλής και πρόεδρο της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων την κυρία Ρουδούλα Ζήση από τον πρόεδρο τη Διαρκού Επιτροπή Εθνική Άμυνα και Εξωτερικών Υποθέσεων, τον κύριο Κωνσταντίνο Βρετό, την πρόεδρο τη Διαρκού Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων, την κυρία Βάσου Παπανδρέου, τον εισηγητή από την κοινοβουλευτική ομάδα του Πασό, κύριο Δημήτρη Ανδρουλάκη, τον εισηγητή από την κοινοβουλευτική ομάδα τη Νέα Δημοκρατία, κύριο Πάνο Παναγιοτόπουλο, από την ε, κοινοβουλευτική ομάδα του Κομμουνιστικού Κόμματο τη Ελλάδα δεν θα παραστεί κάποιο εκπρόσωπο, από τον εισηγητή από την κοινοβουλευτική ομάδα του Λάου, κύριο Κωνσταντίνο Ιβαλιώτη, από τον εισηγητή από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ του κ. Δημήτρη Παπαδημούλη και θα κλείσει η συνεδρίαση με σύντομη δευτερολογία του κ. Σούλτς. Θα παρακολούσα τώρα την κυρία Ροδούλα Ζήση να πάρει το λόγο, ε, καλύτερα από κάτω, γιατί είναι τρίλεπτη. Και παρακαλώ να μείνουμε στο τρίλεπτο, γιατί το πρόγραμμα είναι πολύ συγκεκριμένο και η υποχρέωση επίση του κ. Σούλτ είναι πάρα πολύ συγκεκριμένε. Παρακαλώ λοιπόν για τρία λεπτά, κυρία Ζήση, και αυτό ισχύει για όλου. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σας καλωσορίζουμε στη Βουλή των Ελλήνων και εκ μέρους Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. Ευχαριστώ θερμά, ευχαριστούμε όλοι θερμά για τον εμπνευσμένο λόγο σας και για το πολύ θετικό μήνυμα που δώσατε. Γνωρίζουμε την προσωπική σας προσήλωση στα ιδανικά της κοινωνικής δικαιοσύνης, της αλληλεγγύης και της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, τα οποία συμμεριζόμαστε είναι μια ευκαιρία σήμερα να συζητήσουμε θεσμικά για το ποια Ευρώπη θέλουμε, όπως αναφερθήκατε, και σε ποια Ευρώπη τελικά θέλουμε να συμμετάσχουμε. Κύριε Πρόεδρε, η κρίση μας έδειξε και μας δίδαξε ότι η Ευρώπη χρειάζεται επιγόντως μια αξιόπιστη και αποτελεσματική οικονομική διακυβέρνηση Ωστόσο, αναπόσπαστο τμήμα αυτής της οικονομικής διακυβέρνησης οφείλει να είναι όχι μόνο οι κανόνες για τη δημοσιονομική πειθαρχία και εποπτεία, αλλά να υπάρξει και μια δικαιοσύνη τελικά στον και ρύθμιση του χρηματοπιστωτικού τομέα, να μιλήσουμε δηλαδή για την αναδιανομή του πλούτου στην Ευρώπη, για την ανάπτυξη, για την απασχόληση. Οφείλουμε να δώσουμε νέα όθηση σε προτάσεις, και εδώ είναι το ερώτημά μου γιατί έχουν αργήσει αυτά να γίνουν, έκδοσης ευρωμολόγων χρέους. Μια ιδέα που βρίσκεται επίσημα στο τραπέζι της δημόσιας διαβούλευσης. Να ελοκληρώσουμε την προσπάθεια για τη θέσπιση ευρωπαϊκής φορολόγησης των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Μιας πρωτοβουλίας που επίσης είναι πάγιο αίτημα του Ελληνικού Κοινοβουλίου, όπως και επιτυχία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα ήθελα λοιπόν και παρακαλώ επιτρέψτε μου να σας επευθύνω την εξής ερώτηση. Ποια είναι η προσωπική σας εκτίμηση κύριε Πρόεδρε για την προοπτική σύντομης θεσμοθέτησης πρώτον ενός ευρωπαϊκού οίκου αξιολόγησης, δεύτερον των κοινών ευρωπαϊκών ομολόγων χρέους και τρίτον της φορολόγησης των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Και βεβαίως ποια είναι η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πάνω στο νέο Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Σύμφωνο. Κύριε Πρόεδρε, έχετε τοποθετηθεί για την οικονομική διακυβέρνηση και μάλιστα για δημοκρατική νομιμοποίησή της. Η Βουλή των Ελλήνων, πρέπει να σας πω ότι έχει θεσπίσει, έχει συγκροτήσει μια υποεπιτροπή στην Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για την Ευρωπαϊκή Οικονομική Διακυβέρνηση. Θα ήθελα λοιπόν ε, να θέσω τα, τα εξή ερωτήματα. Ποιες θα είναι οι ε, οι πρωτοβουλίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ενίσχυση της δημοκρατικής εποπτείας της ευρωπαϊκής οικονομικής διακυβέρνησης. Με ποιους τρόπους θα διεκδικήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την καταπροτεραιότητα εφαρμογή των αναπτυξιακών πτυχών της στρατηγικής Ευρώπη 2020 πώς σκοπεύει το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο να προωθήσει μια δικαιότερη κοινωνική αναπτυξιακή στρατηγική ώστε να αμβληθούν οι ανισότητες, η ανεργία και οι αποκλεισμοί που απειλούν την ευρωπαϊκή κοινωνική συνοχή. Τέλος, θα ήθελα κύριε Πρόεδρε να θυμίσω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων έχουν συμμετάσχει πολλές φορές στα διεθνή φόρα και κυρίως στην ΚΟΖΑΚ. Θέλουμε λοιπόν μια δημοκρατική συνεργασία πάνω σε θεσμικές βάσεις. Η ενίσχυση της ΚΟΖΑΚ με συγκεκριμένο ρόλο και δυνατότητες παρέμβασης και διεκδίκησης ενώπιον των ευρωπαϊκών θεσμών είναι μια κίνηση απαραίτητη προς αυτή την κατεύθυνση. Κύριε Ζήση, παρακαλώ να ολοκληρώσετε. Ολοκληρώνω κύριε Πρόεδρε. Ε, ε, λέγοντας ότι θα επιθυμούσα να ακούσω ε, τις δικές σας απόψεις πάνω στους τρόπους με τους οποίους μπορεί να επιδιωχθεί η εντατικοποίηση του πολιτικού διαλόγου μεταξύ του Ευρωπαϊκού και των Εθνικών Κοινοβουλίων και η θεσμοθέτηση συντονισμένης πολιτικής δράσης. Εμείς πιστεύουμε πραγματικά στην Ευρώπη των λαών και σε μια τέτοια Ευρώπη η Ελλάδα αναλαμβάνοντας το μερίδιο της ευθύνης που της αναλογεί και με τις μεγάλες θυσίες και την αποφασιστικότητα του λαού της που επιθυμεί την πρόοδο, τη δικαιοσύνη και την προκοπή θα είναι σε θέση να διεκδικήσει ισότιμα τη δική της προοπτική. Εσείς είστε Έλληνες όπως λένε όλοι οι Ευρωπαίοι και εμείς είμαστε Ευρωπαίοι κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ. Τον λόγο έχει ο πρόεδρος Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, κ. Κωνσταντίνος Βρετός. Επίσης για τρία λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Σούτσα, εκ μέρου των μελών της Επιτροπής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας και για την ομιλία σας και ιδιαίτερα για τα καλά λόγια που είπατε για τον ελληνικό λαό. Πρώτον, ε, επειδή ξέρω, μιλάω σαν έναν έμπειρο πολιτικό, έχετε ξεκινήσει από καλός επαγγελματίας, σαν εκδότης, στη συνέχεια γίνεται δημοτικό σύμβουλο και ανεβήκατε σιγά σιγά αλλά σταθερά την ιεραρχία τη πολιτική ε, της, στην, στη χώρα σα. Ξέρω ότι αυτά που είπατε για τη χώρα μας τα εννοείτε. Και ότι αυτά που προτείνατε επίσης τα εννοείτε. Και ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Τώρα, ε, εμεί σαν πολιτικό σύστημα στη χώρα μας αναγνωρίζουμε τις ευθύνε μας για τα λάθη που κάναμε και τις παραλήψεις που κάναμε στο παρελθόν ώστε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο που φτάσαμε. Πέρα από αυτό όμω υπάρχουν και άλλες ευθύνες οι οποίες είναι έξω από τη δική μας σφαίρα. Και μιλάω πιο συγκεκριμένα για τι ευθύνε της Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία χρόνια σε σχέση με την ελληνική κρίση, που δεν είναι ελληνική κρίση. Είναι ευρωπαϊκή κρίση και θα πρέπει να το προσέξουμε πάρα πολύ. Δεν κινδυνεύει μόνο η Ελλάδα, κινδυνεύουν και άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ακόμα και αυτές που υποτίθεται είναι δυνατέ. Ε, άρα λοιπόν είναι, είναι συλλογικό θέμα και δεν αφορά μόνο τη, μόνο τη χώρα μα. Ε, είπατε ότι είναι επικραμμένοι οι Έλληνε και γυρίζουν την πλάτη στην Ευρώπη. Δεν την γυρίζουν οι Έλληνε την πλάτη στην Ευρώπη. Όχι. Αν ρωτήσετε του Έλληνε και του ρωτάμε, το 75-80% είναι υπέρ τη Ευρωπαϊκή Ένωση ακόμα και τώρα που είναι επικραμμένοι. Είναι υπέρ τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Μερικέ φορέ όμω ορισμένοι Ευρωπαίοι συναδελφοί μα γυρίζουν αυτή την πλάτη στου Έλληνε και λένε ότι είναι αυτή η Ευρώπη. Αυτό πρέπει να το προσέξουμε κύριε, κύριε Πρόεδρε πάρα, πάρα πολύ. Αναγνωρίζουμε ότι υπάρχει το πολιτικό κόστος και σε συναδέλφους μας στα άλλα κοινοβούλια. Και καταλαβαίνουμε ότι θα πρέπει να αιτιολογήσουν την ψήφο τους, αλλά να μην ξεπερνούν τα όρια ορισμένοι από αυτούς, γιατί πράγματι ορισμένοι από αυτούς τα ξεπέρασαν τα όρια και μίλησαν με απρεπή τρόπο για το σύνολο του ελληνικού λαού. Είναι κάτι που δεν μας ταιριάζει, δεν μας αρμόζει, δεν μας πρέπει και εσείς ο ίδιος είπατε πόσο έχετε μεγάλη, σε μεγάλη υπόλοιψη Τώρα, τελειώνοντα κύριε Πρόεδρε, να πω ότι υπάρχει ένα δημοκρατικό έλλειμμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το δείχνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα όργανα τη εκτό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το Συμβούλιο Υπουργών, τα, τα Συμβούλια Υπουργών, τα Συμβούλια Κορυφή, η, η Επιτροπή. Από ό,τι φαίνεται κυδαιμονεύονται από τα κράτη που είναι ψηλά. Με λίγα λόγια, τα ορισμένα κράτη αποφασίζουν και τα όργανα τη Ευρωπαϊκή Ένωση πειθαρχούν πλην και αυτό είναι πολύ παρήγορο, ε, παρήγορο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Άρα λοιπόν θα πρέπει να τονώσουμε, είναι ευκαιρία τώρα κύριε Πρόεδρε, να τονωθεί ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σε αυτή την κρίση, όχι της Ελλάδας, αλλά της Ευρώπης, να, πάρετε πρωτοβουλίες ιδιαίτερες, ώστε η φωνή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να ακουστεί και στην πράξη. Και κατά επέκταση, ο, η συνεργασία των Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τα, με τα Ελληνικά Κοινοβούλια να μεγαλώσει. Να γίνει δηλαδή ένας μια αναδιάταξη των σχέσεων ανάμεσα στα εθνικά κοινοβούλια και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό θα πρέπει κατά την άποψή μου να είναι ένας από τους μεγάλους στόχους σας. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Το λόγο έχει η Πρόεδρος Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων, η κυρία Βάσου Παπανδρέου. Ε, κύριε Πρόεδρε, χαίρομαι που είστε πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και χαίρομαι που είστε εδώ και πιστεύω ότι με εσάς πρόεδρο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα, μέσα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του θα είναι πιο δυναμικό και πιο αποτελεσματικό και το χρειαζόμαστε ειδικά αυτή την περίοδο. Όπως γνωρίζετε ήμουν επίτροπος πριν από πάρα πολλά χρόνια, τότε ήμουν υπεύθυνη για τα κοινωνικά δικαιώματα, τις κοινωνικές υποθέσεις και μαζί με τον κύριο Ντελόρ είχαμε το κύριο θέμα τη χάρτα των δικαιωμάτων των εργαζομένων και η αντίθεσή μας, μάλλον η αντίδραση ήταν από την κυρία Θάτσερ. Κυρία Θάτσερ όμως οχριά μπροστά στο ότι γίνεται σήμερα. Σήμερα και τότε ποτέ δεν φανταζόμουν ότι σήμερα σαν βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου θα μου επέβαλαν να ψηφίσω κατάργηση βασικών δικαιωμάτων των εργαζομένων και αναρωτιέμαι κύριε Πρόεδρε, εγώ δεν τα ψήφισα, τα ψήφισαν οι υπόλοιποι, αλλά είναι νόμος του κράτους. Τι είδου Ευρώπη βλέπετε όταν μια χώρα η οποία έφτεξε, η οποία έχει κάνει τεράστια λάθη, η οποία πρέπει να πληρώσει, θα είναι μέλος μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς βασικά εργατικά δικαιώματα. Ακολουθείτε μια πολιτική, ας αφήσουμε τα δικά μας τα λάθη, εμείς πληρώνουμε για τα δικά μας τα λάθη, αλλά πληρώνουμε και τα λάθη του ευρώ. Ακολουθείτε μια, ακολουθείτε μια πολιτική στην Ευρώπη που 13 χώρες το 2011 δεν είχαν πιάσει το στόχο του 3% το έλλειμμα. Άρα το δημοσιονομικό πλαίσιο ε, ε, ε, υπέστη πλήγμα στην αξιοπιστία του. Τι θα γίνει, θα πάρουν μέτρα για μεγαλύτερη ύφεση στην Ευρώπη. Ήδη πάμε σε ύφεση στην Ευρώπη. Ποιος είναι ο στόχος της πολιτικής που ακολουθείτε. Το 2008 είμαστε όλοι εναντίον των τραπεζών. Σήμερα τράπεζες κάνουν κουμάντο και στην Ευρώπη και παντού. Μας επιβάλλεται ένα μνημόνιο. Έχουμε κάνει λάθη. Δεν, ε, ε, το αφιτσιτώ αυτό σε καμία περίπτωση και πρέπει να μειωθεί το επίπεδο των Ελλήνων. Αλλά σε επευλήθη με τη δική μας την ανοχή ή την ανικανότητα ένα μνημόνιο που είναι λάθος συνταγή. Και τώρα έχουμε ένα δεύτερο μνημόνιο που είναι μεγαλύτερο λάθος, διότι μας οδηγεί Έχουμε πέντε χρόνια ύφεση στην, ε, στην Ελλάδα και φέτος έχουμε μεγαλύτερη ύφεση από την περσινή που ήταν 7% και αυτό που το πακέτο σωτηρίας είναι πακέτο διάσωσης των τραπεζών. Θα τα βάλουμε τα χρήματα σε έναν ειδικό λογαριασμό για να πληρώνονται οι τράπεζες και οι δανειστές μας και θα δεσμεύσουμε ακόμη και έσοδα του ελληνικού δημοσίου φορολογικά που πρέπει να αυξηθούν, πρέπει να μειωθεί η φοροδιαφυγή ή και τελωνιακά έσοδα για να πληρώνονται πρώτα οι τόκοι και μετά οι συντάξεις. Είναι αυτό, έχει αυτό την αίσθηση δικαίου και μπορεί καμία πολιτική τάξη παρόλο ότι έχει προβλήματα η πολιτική τάξη στην Ελλάδα, όλο το πολιτικό σύστημα είναι κατώτερο των περιστάσεων, μπορεί αυτό το πράγμα να επιβιώσει. Μήπως οδηγείται η χώρα σε καταστροφή και εξαθλίωση η κοινωνία αντί να δώσετε μια ευκαιρία στην Ελλάδα να συνέλθει, να ακολουθήσει μια πολιτική η οποία σιγά σιγά θα ξεπεράσουμε όλες αυτές τις δυσκολίες. Κύριε Πρόεδρε, εγώ πολύ έτσι έχω ε, προβληματισμό γιατί σήμερα έχει πάλι δημιουργηθεί αυτή η απόσταση μεταξύ Βορρά και Νότου που δεν είναι καλό για κανέναν, ούτε για τον Βορρά, ούτε για τον Νότο. Τα δικά μας τα ελλείμματα είναι πλεονάσματα του Βορρά. Εάν δεν υπάρξει μια πολιτική ανάπτυξης όλης της Ευρώπης, πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτή την κρίση. Εκτός και αν και εσείς πιστεύετε, που πιστεύω δεν το πιστεύετε, ότι θα πρέπει τελικά να πληρώσουν οι αυτοί οι οποίοι φταίνε λιγότερο. Γιατί αυτοί που πληρώνουν σήμερα με όλα τα μέτρα και εδώ αλλά και στις άλλες τις χώρες με τα πακέτα λιτότητας είναι συνήθως οι πολίτες που έχουν συμμετάσχει λιγότερο στη σημερινή κρίση. Ενώ αυτοί που είναι υπεύθυνοι... Ολοκληρώστε Ολοκληρώνω κύριε Πρόεδρε, γιατί με, ή σε μεγάλο βαθμό υπεύθυνοι για τη σημερινή κρίση ξανά κάνουν κουμάντο. Εγώ θα ήθελα μια διαφορετική Ευρώπη και προσβλέπω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να παίξει έναν πιο αποτελεσματικό και έναν πιο διεκδικητικό ρόλο γιατί σε λίγο φοβάμαι ότι οι πολίτες όπως είπατε δεν θα είναι και τόσο προευρωπαίοι και αυτό δεν είναι καλό για όλους μας. Το λόγο έχει ο εισηγητής από την ομάδα του Πασό, Δημήτρης Κύριε Πρόεδρε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ε, πρέπει να γνωρίζετε ότι οι Έλληνες στη συντριπτική τους πλειοψηφία είναι υπέρ της Ευρωζώνης, υπέρ του ευρώ, αλλά ωστόσο αισθανόμαστε την ανάγκη ενός νέου ιστορικού συμβιβασμού μεταξύ Βορρά-Νότου, ο οποίος θα θεραπεύει γενετικές ατέλειες του ευρώ που μας έκαναν έξι χρόνια Γερμανού στην άνοδο και τρία, τέσσερα χρόνια Αργεντινού στην κάθοδο στη βάση της εξή συμφωνίας. Εμείς θα μειώσουμε τα δημοσιονομικά μας ελλείμματα ή τα χρέη μας, το οφείλουμε αυτό στα παιδιά μας, όχι στη Μέρκελ όπως νομίζουν ορισμένοι, θα μειώσουμε τα ελλείμματά μας, θα επιταχύνουμε τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, εμείς οι Νότιοι, αλλά οι Βόρειοι πρέπει να μειώσετε τα πλεονάσματά σας αυξάνοντας την εγχώρια ζήτηση στις χώρες σας, αγοράζοντας προϊόντα του Νότου ανακυκλώνοντας με παραγωγικές επενδύσεις τα πλεονάσματά σας στο Νότο. Δηλαδή χρειαζόμαστε μια αναπτυξιακή μεταβίβαση πόρων, ας πούμε αυτό που λένε συμβατικά κακός νέο ευρωπαϊκό σχέδιο Μάρσαλ, δηλαδή ένα νέο ευρωπαϊκό σύμφωνο ανάπτυξης, ανασυγκρότησης, συνοχής. Χωρίς αυτό η νέα δημοσιονομική συνθήκη θα είναι μετέωρη και δεν πρόκειται να θωρακίσει την Ευρωζώνη απέναντι στις σεισμικές δονήσεις της κρίσης. Γιατί να έρθουμε μετά δύο-τρία χρόνια εδώ πάλι να σας ζητάμε ένα τρίτο πακέτο διάσωσης αναπόφευκτο αν συνεχιστεί το σπιράλ ύφεσης χρέους. Γιατί να έρθουμε τα τρία χρόνια να σας ζητάμε 50 δισεκατομμύρια, ξέρω 60 δισεκατομμύρια και δεν βάζουμε τώρα τα μισά σε ένα νέο αναπτυξιακό πακέτο που όπως είπα, που ονομάστηκε Ευρωπαϊκό Σχέδιο Μάρσαλ. Το μέγεθος της εμπλοκής της Ευρωζώνης στη διάσωση της Ελλάδας είναι κολοσσίο. Πλησιάζει τα 480 δισεκατομμύρια. Αυτό δημιουργεί ένα ισχυρό πλέγμα αλληλεξάρτησης το οποίο στην πραγματικότητα, αν βάλουμε τα νούμερα, είναι ένα ατελές βεβαίως, ασύμετρο, αλλά de facto ευρωομόλογο. Γιατί δεν κάνουμε το πραγματικό τότε ευρωομόλογο και αν εν πάση περιπτώσει υπάρχουν αντιδράσεις από τις χώρες του πυρήνα της Ευρωζώνης γιατί δεν προχωρούμε σε ένα πραγματικά γενικευμένο αναπτυξιακό ευρωομόλογο αναπτυξιακού σκοπού για να στηρίξουμε αυτό το ευρωπαϊκό σχέδιο Marshall, να μαζέψουμε χρήματα από τι αγορέ. Εμεί δεν θέλουμε τα χρήματα των φορολογουμένων τη Ευρώπη. σα ίσα το Marshall θα είναι προάγγελο για μια μαζική είσοδο κεφαλαίων στη χώρα μα, η οποία θα ευθυγραμμίζεται με ένα εθνικό σχέδιο ανάπτυξη και ανασυγκρότησης. Αυτό το ζήτημα σας βάζουμε. Αυτό που είπατε για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, μην αστευόμαστε. Είναι μηδαμινά ποσά. Εδώ χρειαζόμαστε ένα επενδυτικό boom. Αυτά που λέει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είναι ψηλολόγια. Είναι ε, στραγάλια όπω λέμε στην Ελλάδα. Χρειαζόμαστε ένα επενδυτικό boom. Και να είστε βέβαιοι ότι εμεί πιστεύουμε στον εαυτό μα ότι θα τα καταφέρουμε. Έχουμε τον πατριωτισμό του Made in Greece. Είμαστε βέβαιοι ότι σε 10 χρόνια, εάν κάνουμε αυτά που λέμε, μπορεί να έχουμε 500.000 νέες θέσεις εργασίας, να αυξήσουμε κατά 20 με 30% την παραγωγικότητα της εργασίας στην Ελλάδα και να βρεθούμε στην 30η θέση στην ανταγωνιστικότητα από την 90 θέση που είμαστε σήμερα. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει από την της Νέας Δημοκρατίας ο κ. Πάνος Κύριε Πρόεδρε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, από την πλευρά της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας σας καλωσορίζουμε και εμείς με αισθήματα φιλίας, σεβασμού και εκτίμησης προς το πρόσωπό σας. Τα αισθήματά μας αυτά ενεργοποιούνται από την αξιολόγηση των πράξεων, των δηλώσεων και των θέσεών σας που αφορούν δύο επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο είναι η ευρωπαϊκή σας δραστηριότητα και το δεύτερο επίπεδο η δραστηριότητά σας στις διμερείς σχέσεις Ελλάδας και Γερμανίας. Η δραστηριότητά σας σε ευρωπαϊκό επίπεδο είχε ένα ακόμη δείγμα. Την ομιλία σας στην αίθουσα της Γερουσίας του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Από το δείγμα αυτό προκύπτει για μία ακόμη φορά ότι επιμένετε σε θέσεις με τις οποίες επιστρέφει ο πολιτικός διάλογος στην Ευρώπη στο βάθρο των θεμελιακών αξιών πάνω στις οποίες βασίστηκε η ευρωπαϊκή ιδέα και το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Γιατί αποτελεί ντροπή κύριε Πρόεδρε για τη σημερινή Ευρώπη να εμφανίζεται θεραπενίδα, παρακολούθημα, εργαλείο και εξάρτηση μιας θεολογίας και μιας μεταφυσικής των αγορών. Αποτελεί ντροπή για τη σημερινή Ευρώπη να υποκαθίσταται ο διάλογος και να υποκαθίστανται τα οράματα του Σουμάν, του Αντενάουερ, του Έρχαρτ, του Σμιτ, του Μπραντ, του Κολ, του Σιράκ, του Μιτεράν με την πιο χιδαία αργό των γιάπης των χρηματιστηριακών αγορών. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Και αποτελεί ντροπή για τη σημερινή Ευρώπη να σύρεται πίσω από μια μεταφυσική και μια θεολογία των αγορών πρωτοφανή για την ευρωπαϊκή ιστορία η μάχη που δίνεται για την Ελλάδα σήμερα εσείς και άλλες πολιτικές προσωπικότητες στον ευρωπαϊκό κόσμο είναι μάχη για την Ευρώπη και όχι μάχη για την προστασία των κοινωνικών και πολιτικών δικαιωμάτων των Ελλήνων. Σε ό,τι αφορά τις διμερείς μας σχέσεις, χαιρόμαστε ιδιαίτερα γιατί με τα όσα λέτε και την εν γέννη δραστηριότητά σας συμβάλλετε αποφασιστικά στο να αποκατασταθεί η σωστή εικόνα της Γερμανίας, του γερμανικού έθνους και της γερμανικής κοινωνίας στην ελληνική κοινή γνώμη. Λυπούμεθα κύριε Πρόεδρε, γιατί υπάρχουν συνάδελφοί σας πολιτικοί, ενεργοί πολιτικοί στη Γερμανία και υπάρχουν και μέσα μαζικής επικοινωνίας στη Γερμανία που τοποθετούνται με τρόπο που προσβάλλει την αξιοπρέπεια του ελληνικού έθνους και την αξιοπρέπεια της ελληνικής κοινωνίας. Όλοι αυτοί είναι δέσμοι ενός πρωτοφανού σε αναχρονισμό γερμανικού επαρχιωτισμού που θίγει την εικόνα της σημερινής Γερμανίας στην Ευρώπη και τον κόσμο. Ομολογούμε κύριε Πρόεδρε ότι και λάθη έκανε ο ελληνικός λαός και καθυστερήσεις υπήρξαν και τεράστια ασφάλματα του πολιτικού συστήματος. Σήμερα όμως ο ελληνικός λαός υποβάλλεται σε βαρύτατες θυσίες που συνεπάγονται τεράστιο πόνο. Γι' αυτό ο ελληνικός λαός αξίζει σεβασμό, ενίσχυση της δικής του αξιοπρέπειας και της διεθνούς του εικόνας και όχι προσβολές και ταπεινώσεις. Κύριε Πρόεδρε, αφού σας ευχαριστήσω για τη σημερινή δημόσια τοποθέτησή σας, θέλω να σας παρακαλέσω τα λόγια που είπατε για την ανάπτυξη να συμβάλλετε για να γίνουν πράξη. Πριν από λίγες μέρες, η μεγάλη πλειοψηφία του Ελληνικού Κοινοβουλίου μπροστά στο δίλημα βεβαία χρεοκοπία ή ρίσκο για τη σωτηρία του τόπου έκανε τη δεύτερη επιλογή. Πήραμε το ρίσκο για να στηρίξουμε τη σωτηρία του τόπου. Αυτό το ρίσκο όμως θα αποδειχθεί άλμα στο κενό για όλους μας, συμπαρασύροντας και το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, αν πολιτικοί του δικού σας κύρους και του δικού σας βεληνεκούς δεν προτάξουν το θέμα της ανάπτυξης μαζί με την ανάγκη των διαθροτικών αλλαγών και της δημοσιονομικής πειθαρχίας. Ευχαριστούμε και πάλι για τη διαρκή σας παρουσία στα θέματα που αφορούν και την Ευρώπη και την Ελλάδα. Τον ε, λόγο έχει από την κοινοβουλευτική ομάδα του λαού ο κ. Κωνσταντιών Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλωσορίζω τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εκ μέρου του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού στη Βουλή των Ελλήνων και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά εκ μέρου του Προέδρου του Λαός, του κ. Καρατζαφέρη, για την ανταπόκριση που δείξατε στην επιστολή που σας έστειλε σχετικά με την κρίση στην Ελλάδα, το ρόλο της Τρόικας και τη συμβατότητα του νέου μνημονίου με το κοινοτικό κεκτημένο. Έχουμε συνεπάρξει, κύριε Πρόεδρε, χρόνια στι Βρυξέλλε, εσείς ω δραστήριο ευρωβουλευτής και εγώ συνεργάτης τεσσάρων ε, Ελλήνων Ευρωβουλευτών τριών διαφορετικών ελληνικών κομμάτων εκπροσωπείται το μόνο δημοκρατικά εκλεγμένο όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το μόνο θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του οποίου τα μέλη εκλέγονται με άμεση και καθολική ψηφοφορία. Σε αυτό το όργανο φτάνει λοιπόν, προσεγγίζει η φωνή των λαών της Ευρώπης κατεξοχήν ταλαιπωρημένος λαός της Ευρώπης είναι ο ελληνικός. Όχι μόνο λόγω της οικονομικής κρίσης που βιώνουμε όλοι, αλλά και λόγω της λαθρομετανάστευσης. Η Ελλάδα, κύριε Πρόεδρε, και οι Έλληνες υποφέρουν από την εφαρμογή του κανονισμού Δουβλίνο 2. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω θερμά να μεταφέρετε στους λαούς της Ευρώπης την αγωνία των Ελλήνων και την επιθυμία τους για την κατάργηση του κανονισμού Δουβλίνο 2 ε, ενός κανονισμού που έχει καταδικάσει την Ελλάδα στην ανεργία και την εγκληματικότητα, σημαντικό μέρος των οποίων, ανεργίας και εγκληματικότητας, οφείλεται στους λαθρομετανάστες. Αναφερθήκατε επίσης κύριε Πρόεδρε στα δεινά που επεσόρευσε ο ναζισμός στην Ελλάδα. Και έτσι ακριβώς είναι. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω, ως σημαίνουσα προσωπικότητα της γερμανικής πολιτικής ζωής, να φέρετε στο προσκήνιο του δημοσίου διαλόγου της χώρας σας το ζήτημα των γερμανικών πολεμικών αποζημιώσεων, των αποζημιώσεων δηλαδή που οφείλει η Γερμανία προς την Ελλάδα, αποζημιώσεις που έχει επισήμως αναγνωρίσει με δήλωση του αείμνης του Έρχαρτ το 1964. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει από την κοινοβουλευτική του ΣΥΡΙΖΑ του συνασπισμού της Ριζοσπαστικής Αριστεράς για τους μεταφραστές. Κύριε Παπαδημούλη για τη ΣΥΡΙΖΑ σκέτους να μην αντιληφθεί πρόεδρος τι σημαίνει ο κ. Δημήτρης Παπαδημούλης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Σούλτς, σας καλωσορίζω και εγώ με τη σειρά μου. Είχα την ευκαιρία στην προηγούμενη θητεία του Ευρωκοινοβουλίου να σας γνωρίσω και να συνεπάρξουμε. Είστε ένας πετυχημένος Ευρωβουλευτής και είναι θετικό γεγονός ότι αναλάβατε πρόσφατα το τιμόνι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αλλά δυστυχώς το τιμόνι της Ευρωζώνης το κρατάει η Αγγέλα Μέρκελ. Είναι αλήθεια ότι ο ελληνικός λαός υποφέρει πολύ, καταβάλει τεράστιο κόστος γιατί πληρώνει αμαρτίες δεκαετιών πολλών ελληνικών κυβερνήσεων. Αλλά πληρώνει και τη δογματική αιμονή σε μια επικίνδυνα λαθασμένη πολιτική της ευρωπαϊκής ελίτ η Ευρώπη που διαφεντεύει η κυρία Μέρκελ δεν είναι η Ευρωπαϊκή Γερμανία του Σμιτ, του Μπραντ, του Σρέντερ, του Κόλ. Είναι το όραμα μιας γερμανικής Ευρώπης που προσπαθεί να βάλει τα πάντα και τους πάντες στο στενό παπούτσι ενός δογματικού νεοφιλελευθερισμού και ενός οικονομικού εθνικισμού. Και αυτό παράγει το ηφαισιακό σπιράλ του θανάτου. Εδρεώνει την κυριαρχία ενός καπιταλισμού καζίνο που ξυλώνει κάθε έννοια και κατάκτηση της ευρωπαϊκής κοινωνικής Ευρώπης. Αυτά που συμβαίνουν σήμερα στην Ελλάδα απειλούν και τους άλλους ευρωπαϊκούς λαούς. Είναι ο γερμανικός τύπος που γράφει ότι με το τελευταίο πακέτο η Ελλάδα μετατρέπεται στην πρώτη απικία της Ευρωζώνης. Πώς είναι δυνατόν να υπάρξει η ανάπτυξη και η δικαιοσύνη για την οποία μας μιλήσατε στο λόγο σας, όταν ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός είναι λιγότερο από 1% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ, όταν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν έχει τη δύναμη που έχει η Αμερικάνικη, η Εγγλέζικη, η Ιαπωνέζικη στο να διαχειριστεί το ευρωπαϊκό χρέος ή να υπερασπίσει το νόμισμα. Όταν δεν υπάρχουν οι μηχανισμοί αναδιανομής και ανακύκλωσης των πλεονασμάτων του Βορρά στο βωμό της συνοχής, της κοινωνικής, της εδαφικής, της περιφερειακής. Τα δύο τρίτα των γερμανικών εξαγωγών ξέρετε πολύ καλά ότι υπάρχουν γιατί είναι εισαγωγές και ελλείμματα και χρέη του Ευρωπαϊκού Νότου. Αν δεν αλλάξουν λοιπόν τα πράγματα στην Ευρώπη με αύξηση του προϋπολογισμού, με αύξηση των πολιτικών συνοχής με ενίσχυση των αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, με ευρωομόλογο, με ευρωπαϊκή διαχείριση του χρέους, τότε η ύφεση, η μεγάλη ανεργία, η μεγάλη μείωση των αποδοχών και των δικαιωμάτων μισθωτών και συνταξιούχων, η αποδόμηση του κοινωνικού κράτους από ελληνικός πόνος θα γίνει ευρωπαϊκό υπόδειγμα. Θα, θα περίμενα λοιπόν, αντί να υπερασπίζεστε αυτό το πρόγραμμα που είναι με πατέντα Μέρκελ να τονίσετε εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τις δικές σας προτάσεις, τις δικές σας απαιτήσει που θέλουν να σπάσουν και πρέπει να σπάσουν το ταχύτερο δυνατό αυτό το φαύλο κύκλο. Γιατί αν σπάσει ο αδύνατος κρίκος της Ευρωζώνης που λέγεται Ελλάδα, τότε θα σπάσει όλη η αλυσίδα και το κοινωνικό και οικονομικό κόστος για όλη την Ευρώπη θα είναι τρομακτικό οι βαθύτατες διαιρέσεις που παράγει αυτή η ανόητη και επικίνδυνη πολιτική τροφοδοτούν ανισότητες κοινωνικές αλλά και την αναβίωση ενός εθνικισμού. 50-60 χρόνια μετά το τέλος του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου όσοι θέλουν μια Ευρώπη πρέπει να αγωνιστούν διαφορετικοί, πρέπει να αγωνιστούν για αλλαγές και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Αλλιώς τα πράγματα θα πάνε προς τα πίσω. Ευχαριστούμε όλους τους ε, συναδέλφους ομιλητές και τη συνεδρία θα κλείσει τώρα με την για ένα δεκάλεπτο δευτερολογία του ο κύριος Μάρτιν Σούλτς. Κύριε Σούλτς έχετε το λόγο. Vielen Dank. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς θα äh, ήθελα να σας ευχαριστήσω για τα σχόλιά σας. Ε, αλλά είμαι σε μια κάπως äh, δύσκολη äh, κατάσταση διότι θα πρέπει να συνδυάσω δύο αποστολές. Είμαι καταρχάς εδώ ως ε, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με μια διπλωματική εντολή ε, και πολλά τα äh, οποία είπατε εμένα με οδηγούν στο μέσο των συζητήσεων του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Ε, εγώ αισθάνομαι μια χαρά γιατί έχω äh, ζήσει ως κοινοβουλευτικός και ξέρω γιατί γίνονται αυτές οι ασκήσεις αλλά θα επιτρέψω να σας απαντήσω με πλήρη ειλικρίνεια η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης χαρακτηρίζεται από τις πλειοψηφίες οι οποίες υπάρχουν στην Ευρώπη. Εγώ αυτό δεν μπορώ να το σχολιάσω αυτό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι η ρεαλιστική ε, πραγματικότητα. Και γι' αυτό το λόγο δεν έχει νόημα να κάνει κανείς κάποια σχόλια. Και εγώ δεν θέλω να κάνω, γιατί εγώ ε, το έχω κάνει στο παρελθόν πολλαπλώ. Αλλά είμαι πρόεδρο ενό θεσμού και πρέπει να σα πω ότι οι αποφάσει οι οποίε παίρνονται στη Σύνοδο κορυφή, στο Συμβούλιο Κορυφή, παίρνονται ομοφόνο. Είναι όλε οι κυβερνήσει παρούσε. Και μετά δεν μπορεί να πει κανεί ότι είναι η Αγγέλα Μέρκελ η οποία διοικεί την Ευρώπη έτσι απλά. Κύριε Σταμού, λυπάμαι, πρέπει να διαμαρτυρηθώ προκειμένου. Διότι εγώ, εδώ και τώρα, και πρέπει να το πω, ε, εγώ να υπεραμηθώ τη Αγγέλα Μέρκελ, δηλαδή για έναν Γερμανό σοσιαλδημοκράτη, αυτό είναι μια άσκηση παραλογισμού. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι η πραγματικότητα. Η Αγγέλα Μέρκελ είναι ένα κομμάτι του Συμβουλίου. Είναι και αυτή η κομμάτι. Αλλά υπάρχουν άλλοι 26 εκεί πέρα. Οι οποίοι όλοι είπανε ομοφόνος ναι ή όχι στα συγκεκριμένα μέτρα. Τώρα, αν αυτά τα μέτρα είναι καλά ή κακά, σωστά ή όχι, αυτό είναι μια συζήτηση η οποία συνεχίζεται. Και ξέρετε, είναι μια συζήτηση όχι μόνο μεταξύ δεξιάς και αριστεράς, είναι και μεταξύ κρατών. Ε, και ομάδων προκειμένου. Είμαστε ειλικρινεί. Και ομάδες και κράτη ομάδων ε, τα οποία είναι, έχουν πολλές διαφορετικές κυβερνήσεις. Δεν είναι δηλαδή ότι στα ευρωπαϊκά κόμματα όλοι είναι υπέρ της μίας ή της άλλης θέσης. Και οι χριστιανοδημοκράτες και οι συντηρητικοί και οι φιλελεύθεροι ε, και στους σοσιαλιστές υπάρχουν πάρα πολλές ετερογενείς θέσεις και απόψεις. Και αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να να προσμετρηθεί έτσι εύκολα αριστερά-δεξιά όπως το ξέρουμε στα εθνικά κοινοβούλια. Η Ευρώπη έχει και μια θεσμική λογική στα πλαίσια της οποίας υπάρχουν και τα ενδιαφέροντα των μεμονωμένων κρατών. Και εδώ ακριβώς είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα τα οποία έχουμε. Ε, πρέπει να βρούμε μια κοινή και κοινοτική μέθοδο, όπως το λέμε εμείς στην Ευρώπη, το οποίο σημαίνει ότι θα πρέπει η μεταφορά των διαφόρων ε, συμφερόντων και ενδιαφερόντων να τα μεταφέρουμε και να τα αντικαθρεπτήσουμε σε επίπεδο κοινοτικών θεσμικών φορών όπου υπάρχουν τα μεγάλα και τα μικρά κράτη και να υπάρχει μια ισορροπία, ένα ισοσκελισμός ενδιαφερόντων μεταξύ μεγάλων και μικρών. Για δεκαετίες η Ευρώπη αυτό το επέτυχε. Από τη στιγμή που υπάρχει η συνθήκη της Λισαβόνας στο Συμβούλιο ε, ξαφνικά υπήρξαν άμεσες αντιπαραθέσεις μεταξύ κρατών. Το οποίο χωρίς αμφιβολία ε, έρχεται και ο τύπος ο οποίος το υποδαβλίζει, οργανώνει, υποστηρίζει. Γι' αυτό όταν μιλάμε στις Βρυξέλλες για την κοινοτική μέθοδο, μιλάμε για μια αλλαγή αυτής αρθέζεται της υφέρπουσας αλλαγής την οποία παρατηρούμε. Ότι ξαφνικά ε, η εξισορρόπηση των ε, μενομενωμένων ενδιαφερόντων ξαφνικά εμφανίζονται ομάδες κρατών ε, τα οποία υπεραμείνονται ενός πακέτου ενώ κάποιοι άλλοι ενός άλλου. Και ξαφνικά ο ένας τραβάει το χαλί κάτω από τον άλλο. Και αυτό είναι ένας λαθασμένος τρόπος. Και εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αυτό το λέμε ότι αυτό πρέπει να το σταματήσουμε και θα πρέπει να ξαναδώσουμε την προ πρωτοπορία στην ευρωπαϊκή μέθοδο. Να μπορέσουμε δηλαδή όλοι μαζί. Κύριε Παναγιωτόπουλο, ελπίζω να το είπα κάπως σωστά. Κύριε Παναγιωτόπουλο, το είπατε γερμανικά πολύ ωραία, λέει ο Πρόεδρος, αλλά το καταλάβαμε τι εννοούσατε ή ποιον εννοούσατε. Λοιπόν, ο εκπρόσωπο τη Νέα Δημοκρατία, εν πάση λέει ο κύριο ο πρόεδρος. Θα ήθελα να σα πω κάτι και να ε, αντιπαρατεθώ λίγο. Έχετε δίκιο σε ένα σημείο. Ναι, στη Γερμανία υπάρχουν ε, ε, εφημερίδες οι οποίες γράφουν τραγικά πράγματα για την Ελλάδα. Ωραία. Και αυτό το ξέρω και εγώ το απορρίπτω. Και έχω προσπαθήσει και στα πλαίσια της ομιλίας μου ότι οι ομαδοποιήσεις, οι ομεγενοποιήσεις, αυτά τα κλισέ υπέρ κατά κρατών και να λέμε ότι το ένα κράτος είναι με, χαρακτηρίζεται από το ένα στερεότυπο πολιτική την οποία χρειαζόμαστε. Αλλά ξέρετε αυτό ισχύει και για την Ελλάδα. Και εδώ γίνεται αυτό. Δεν το βρίσκω καλό ότι η κυρία Μέρκελ, συγγνώμη, είναι η, η πρωθυπουργό η οποία ξέρει χθε στο Bundestag με τη δικό μου το κόμμα στο οποίο εγώ ανήκω, είμαι σοσιαλιστή, με όλα τα äh, κόμματα, με του πράσινου, με ένα μεγάλο μέρο των φιλελευθέρων. Ήταν υπέρ ενό σωσιβίου για την Ελλάδα, ενό πακέτου βοηθεία. Ξαφνικά εδώ λέτε ότι είναι ε, ε, ένας αξιωματικός στο να ζει και έτσι να παρουσιάζεται. Είναι απαράδεκτο, πρέπει να σας το πω. Ε, λοιπόν, συγγνώμη, το ίδιο ισχύει και για τον κύριο Σόιμπλε και για άλλους πολιτικούς. Και εσείς κάτι τέτοιο κάνετε. Λοιπόν, αυτό το οποίο θα πρέπει να ξέρουμε όλοι είναι κάτι διαφορετικό. Όταν είμαστε στην Ευρώπη και βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου το οικονομικό και το νομισματικό πρόβλημα το οποίο έχουμε οδηγεί ώστε να ξανααναφύονται όλα τα παλιά στερεότυπα και όχι μόνο αυτά αλλά να υπεραμεινόμεθα και αυτόν τότε όλοι εμείς και εσείς στην Ελλάδα, εμείς στη Γερμανία, όλοι εμείς, όλοι θα πρέπει πραγματικά να μας κούρουν σε ένα κόδωνα κινδύνο γιατί αυτό δείχνει ότι τα δαιμόνια του 20ου αιώνος ε, το μίσος, ε, οι γεμονικές τάσεις, η αδιαφορία όσον αφορά τις μειονότητες, ε, ο ένας λαός κατά το άλλο, ότι όλα αυτά τα δαιμόνια είναι ζωντανά στον 21ο αιώνα και μπορούν να αναζωοποιηθούν αν εμείς δεν προσπαθήσουμε να τα ελέγξουμε. Γι' αυτό το λόγο ακριβώς θα πρέπει ο κάθε δημοκράτης πολιτικός τέτοιες εκφάνσεις, τέτοια στερεότυπα και τέτοιες εξελίξεις πραγματικά να τα απορρίπτει και αδράχνομαι τις ευκαιρίες και να το κάνω αυτό όπως βλέπω ότι το κάνατε και εσείς και βλέπω ότι συμφωνείτε με αυτό που λέω. Πρέπει να το κάνουμε όλοι. Χρειαζόμαστε, είτε αυτό το λέμε τώρα πλάνο Marshall ή οτιδήποτε, χρειαζόμαστε επενδύσεις, δεν ξέρω πώς θα το πούμε, αλλά επενδύσεις χρειαζόμαστε. Πρέπει να επαναφέρουμε τους επενδυτές σε αυτή τη χώρα και σε άλλα κράτη. Αλλά ο επενδυτής θα έρθει μόνο εδώ και να βοηθήσει και να επενδύσει ή το κάνει μικρό, μεγάλο, δεν ξέρω σε επίπεδο, μόνο εάν υπάρχει εμπιστοσύνη. Κανένας er άνθρωπος δεν θα βάλει μία δραχμή κάπου αν δεν έχει εμπιστοσύνη. Oh, Κανένα δεν θα πάει να βάλει λεφτά αν έχει την εντύπωση ότι ξέρει θα επενδύσω αλλά. Κανένα δεν θα επενδύσει εάν ε, de facto έχουμε ατέλειωτα γραφειοκρατικά και νομοθετικά εμπόδια, το οποίο όχι θα βοηθήσουν την επένδυση, αλλά θα την κάνουν πιο ακριβή ή πιο δύσκολη. Για αυτούς του λόγου είναι βασική προπόθεση όπω η Ελλάδα δημιουργήσει πάλι εμπιστοσύνη, αποθεματικό εμπιστοσύνη. Και αυτό είναι κάτι το οποίο μπορείτε να το κάνετε μόνο εσεί στην Ελλάδα και μπορείτε να το κάνετε μόνο αν υπάρχει πραγματικά μια μετενέργεια, μπορώ να το πω έτσι, στις ε, αποφάσει και τι αλλαγέ τι οποίε θα περάσουμε σήμερα. Δεν πιστεύω ότι η Ευρώπη μέχρι σήμερα δεν έκανε τίποτα. Είπατε προηγουμένω ε, νομίζω ήταν ο κύριος, νομίζω Ανδρουλάκης, ελπίζω ε, να το λέω σωστά και αυτό. Ε, λοιπόν, είπατε, ε, δεν έχουμε, ακούσαμε πολλά από την Ευρώπη μέχρι σήμερα. Όχι, ακούσατε. Η Ευρώπη έδωσε δισεκατομμύρια τα οποία επέρασε σε εσά. Αυτό όμως το οποίο σαν Ευρωπαίοι πρέπει να καταλάβουμε, δεν αρκεί αυτό να στέλνουμε τα πακέτα των εκατομμύριων και των δισεκατομμυρίων. Αυτό το χρειάζεται αυτή η χώρα είναι επενδύσεις επενδύσει για μελλοντικέ εξελίξει στη βιομηχανία και στην οικονομία. Προσπάθησα να σα πω κάποιε, όπω αν θέλετε η ηλιακή ενέργεια, ε, η αλληλεγγύη με τα κράτη τη Βορείου Αφρικής δεν έχει σημασία. Αλλά όπου και πρέπει να επενδύσει κανεί πάνω από όλους του νέου ανθρώπου αυτού τη χώρα. Αν πραγματικά αποδεχτείτε το γεγονό οτι ότι 30-40 των νέων οι οποίοι ίσω έχουν και πολύ καλέ σπουδέ, μια ολόκληρη γενιά δεν θα βρουν δουλειά, αυτό είναι τραγικό. Γι' αυτό επαναλαμβάνω και το είπα και äh, προηγουμένω. Περιμένω την πραγματικότητα. Ο κύριο Παπαδήμο αύριο με την Κομισιόν να μιλήσει και να διαπραγματευτεί αύριο πώ τα κονδύλια τα οποία δεν έχουν χρησιμοποιηθεί από το κοινωνικό ταμείο, από άλλα ταμεία, να μπουν σε προγράμματα απασχόληση νέων um ανθρώπων, όχι μόνο στην Ελλάδα και σε άλλα κράτη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ήξερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι έτσι ότι εμεί θα πρέπει να τηρήσουμε το χρόνο ομιλία. Θα το κάνω, ξέρετε, και στο Ευρωπαϊκό Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ. Αλλά αυτή την εμπειρία την είχαμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όταν ήρθα εγώ προσκεκλημένο μου κόψαν τον χρόνο. Αλλά άμα θέλετε να πείτε κάτι παραπάνω, εγώ δεν έχω αντίρρηση, λέει ο πρόεδρο Πετσάλικο. Ευχαριστούμε τον ε, κύριο Μάρτιν Σούλτ για την ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα αρχική του τοποθέτηση αλλά και για τις απαντήσεις, η κατάθεση απόψεων που έκανε στην δευτερολογία του και ευχαριστώ επίσης και όλους τους ε, συναδέλφους και τις συναδέλφους που παρευρεθήκατε, πήρατε μέρος σήμερα σε αυτήν την ειδική συνεδρίαση.